η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικής Αφρικής. Ο κύριος Λάγκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πίτροπα, αγαπητοί συνάδελφοι. Με τις αφρικανικές χώρες, τα αφρικανικά κράτη είχαμε μακρές διαπραγματεύσεις για να συνάψουμε συμφωνίες εταιρική σχέσης και να τις διαμορφώσουμε έτσι ώστε να είναι όριμες προς υπογραφή και προς κύρωση, να έρθουν στο Κοινοβούλιο. Εμείς το επιθυμούμε διότι πραγματικά θέλουμε να αναπτυχθούν οικονομικά οι χώρες αυτές της Αφρικής και σε περιφερειακό επίπεδο να ενισχυθεί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Δυτική Αφρική. Πολλές χώρες εξαρτώνται πάρα πολύ από τις εξαγωγές τους και μάλιστα ε, δεν έχουν αναπτύξει το ενδοπεριφερειακό τους εμπόριο και την οικονομία τους. Γι' αυτό έχουμε πολλά ασύμμετρα στοιχεία εκεί έχουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, ε, ε, έχουμε εξαιρέσει από τις συμφωνίες κάποιους ευαίσθητους τομείς για να ενισχυθεί η περιφερειακή προστιθέμενη αξία. Και είναι σαφέστατο αυτό. Αν δούμε τι γίνεται στη Δυτική Αφρική, 80% πούμε ε, των εισαγωγών κακάο όπου ε, εμείς ε, καταναλώνουμε και μόλις 4% της σοκολάτας. Δηλαδή εισάγουμε ε, πρώτη ύλη το κακάο αλλά όχι τη σοκολάτα. Χρειάζεται λοιπόν προστιθέμενη αξία στη μεταποίηση εκεί. Στη Δυτική Αφρική βέβαια τίθενται και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Για να επανέλθω στο κακάο γνωρίζουμε ότι την ε, συλλογή του καρπού, ε, το κακάο, χρησιμοποιούν παιδική εργασία. Και δεν μπορώ να φανταστώ ε, όταν τρώμε σοκολάτα παιδική, τα παιδιά μας τρώνε σοκολάτα, προωθούμε την παιδική εργασία στον κλάδο του κακάου στη Δυτική Αφρική. Γι' αυτό το θέμα της αηφορίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ υπάρχει το εξής περίεργο πράγμα. Ε, έχουμε μία συμφωνία εταιρική που πάνω κάτω λειτουργεί. Τα ξέρει αυτά ο Ντέιβιτ Μάρτιν. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κεφαλογιά την αηφορία, έχουμε πάρα πολύ θετικές αναφορές και πολλές. Και για να το συνδέσω τώρα με την Δυτική Αφρική και το συγκρίνω, κύριε Επίτροπε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Γι' αυτό σας ερωτούμε και κάνουμε αυτή την προφορική ερώτηση. Τι γίνεται με την εφαρμογή ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πώς θα τα εξασφαλίσουμε. Στο Καριφόρουμ υπάρχει ε, σαφής αναφορά στους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταναγκαστική παιδική εργασία. Ε, γίνεται αναφορά ξεχωριστή. Και μια δεύτερη ερώτηση Υπάρχει ένα συμβουλευτικό όργανο εκεί που θα πρέπει λέει να συσταθεί και εκεί λείπει από τη συμφωνία μια ε, σαφής περιγραφή, μια συγγραφή υποχρεώσεων και καθηκόντων ε, και πάλι ε, διαφέρει αυτό με το CAI Forum. Λοιπόν, πώς ορίζονται οι ευθύνες, τι πόρους έχει αυτό το όργανο, πώς λειτουργεί, πώς έχουν οι διαδικασίες, όλα αυτά ορίζονται στη Συμφωνία Καριφόρουμ συμπεριλαμβάνονται τα θέματα του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου. Και τι γίνεται με τη διευθέτηση των διαφορών. Υπάρχουν μηχανισμοί διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφορών. Και στην τρίτη ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται η DigiTrade, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, αλλά και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πώς θα εξασφαλίσουν ότι οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών θα ε, συμπεριληφθούν με τρόπο που τους αρμόζει. Και επίσης θέλουμε να μάθουμε και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα όλων αυτών των υποθέσεων. Έτσι ώστε όταν κάνουμε αυτές τις συμφωνίες και ερχόμαστε να τις εφαρμόσουμε, να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει επαρκή αηφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκε. Κυρία Μάλστρομ. Η Επιτροπή και εγώ η ίδια εξάλλου έχουμε υποβάλει κάποιες προτάσεις και έχουμε κάνει τις ανακοινώσεις μας από πέρσι, ιδιαίτερα τα αποτελέσματα που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη κάτι που πάντα αποτελεί συνιστόσα των συμφωνιών μας. Πρόκειται για κάτι που καταρχήν εμπεριέχεται στην Συμφωνία του Κοτονού. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους στόχους, καθώς βεβαίως και η συνιστόσα, η κοινωνική και η περιβαλλοντολογική. Αναφερόμαστε στα δικαιώματα αυτά, καθώς και στα πρότυπα και για το περιβάλλον, αλλά και για την εργασία, τα πρότυπα του ΑΕΛΟ. Η συμφωνία αυτή εταιρική σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικής Αφρικής συμπεριλαμβάνει αυτές τις πηγές και εμείς θα λάβουμε υπόψη μας και την υλοποίησή της και την παρακολούθηση. Βεβαίως υπάρχει το παρατηρητήριο για την ανταγωνιστικότητα που παρακολουθεί όλες αυτές τις ε, πτυχές αυτής της συμφωνίας κατά την υλοποίησή της. Υπάρχει βεβαίως και το χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για μια ε, συμφωνία η οποία αναθεωρείται και αξιολογείται κάθε πέντε χρόνια. Είναι μακροπρόθεσμη στόχοι και φυσικά αξιολογούνται όλοι οι τομείς. Το περιβάλλον, όπως σας είπα, τα πρότυπα στον τομέα της εργασίας, και βεβαίως κάθε φορά που γίνεται η αναθεώρηση η αξιολόγηση μπορεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα είτε να προταθούν και τροπολογίες και τροποποίηση στην εταιρική αυτή σχέση. Πρέπει οι δύο εταίροι να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, τις υποχρεώσεις τους και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και όσον αφορά την εργασία, τις συνθήκες εργασίας. Και αυτό ισχύει και θα γίνει ξεκινώντας από πολιτικό διάλογο, αλλά και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και την διακοπή, το ίστατο όπλο, αν θέλετε. Έχουμε ήδη λοιπόν ξεκινήσει την προετοιμασία με τις χώρες της Δυτικής Αφρικής για την ε, δημιουργία ενός ε, συμβουλευτικού οργανισμού Προβλέπουμε οικονομική στήριξη για τον φορέα αυτό και για την ε, διαβουλευτική αυτή επιτροπή. Έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε αυτούς τους θεσμούς για την ορθή αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Αυτό μπορεί να γίνει καθώς και η υποβολή κάποιων συστάσεων από μέρους αυτών των οργανισμών τα δύο μέλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάσουν περιπτώσεις μη τήρησης ή παραβίησης των διατάξεων της ε, Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Και εάν χρειάζεται κάτι τέτοιο να υπάρξει και αλλαγή της ε, πολιτικής. Σε όλους τους τομείς η παραβισεις των διαταξεων της εξετάζει και αξιολογεί την επιτευχθήσα πρόοδο σε κάθε περίπτωση θα θέλουμε να υπάρχει συνοχή και εντελεχής έλεγχος της υλοποίησης αυτής. Θα ήταν πολύ καλό αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τώρα αρχίσει να δεσμεύεται έτσι ώστε παραδείγματος χάρη να δημιουργηθεί μια κοινή ε, κοινοβουλευτική επιτροπή με τις χώρες της Δυτικής ε, Αφρικής. Αυτό θα βοηθήσει και θα συνεισφέρει σημαντικά στην ευάθυνση αυτής της ε, πολιτικής συνεργασίας. Και σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον πολιτικό διάλογο αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει και να συνοδεύσει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ του ΕΛΚ, ο κύριος Κάσπαρη έχει 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αν κοιτάξει κανείς τις τελευταίες εβδομάδες και το τελευταίο, τους τελευταίους μήνες από που έρχονται οι περισσότεροι πρόσφυγες βλέπουμε πολλούς από την Αφρική. Η κατάσταση λοιπόν στην Αφρική πρέπει να βελτιωθεί. Οι συνθήκες ζωής και εργασίας αυτών των ανθρώπων πρέπει να βελτιωθούν. Δεν μπορούμε βεβαίως να κάνουμε τα πάντα εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε όμως να συνεισφέρουμε στο βαθμό που μας το επιτρέπει η ε, συμφωνία και οι σχέσεις που έχουμε με τις χώρες αυτές. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα που ήδη ανέφερε ο συνάδελφος Μπέρν Λάγκε. Σίγουρα πρόκειται για μια συμφωνία που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Γιατί έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Καταρχήν, ποιος, πώς ξεκίνησε αυτή η συμφωνία εταιρικής σχέσης. Τι μπορεί λοιπόν στα πλαίσια αυτά να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα στην Δυτική Αφρική υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ορθά αν υπάρχει ένας από τους δύο εταίρους που ελέγχει και επιβάλλει στον άλλο εταίρο. Θα ήταν λοιπόν πολύ καλό να δείξουμε ότι ακούμε αν θέλετε τους ε, εταίρους μας και ότι στηρίζουμε την ε, ε, συμπερίληψη και άλλων κρατών από τη Δυτική Αφρική σε αυτή τη συμφωνία. Η κυρία Κέρτον Ντάρλιν, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πέρσι το φθινόπωρο. κυρία Επίτροπε, μιλήσατε για το εμπόριο για όλους και μας είπατε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και το εμπόριο θα συμβαδίζουν. Σήμερα μιλάμε για μια εμπορική συμφωνία με τη Δυτική Αφρική, όπου δυστυχώς δεν λαμβάνουμε υπόψη τη βιωσιμότητα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι ύψης της σημασίας δεν έχουμε τα μέσα έτσι ώστε τα δικαιώματα αυτά να αποτελέσουν πραγματικότητα και όχι να βρίσκονται στο χαρτί. Αυτό θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη όπως έκανε στις συμφωνίες εμπορίου τα τελευταία δέκα χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαίος εμβασμός, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν οι ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν για τον υπόλοιπο κόσμο. Χρειάζονται βελτιώσεις. Ο κύριος Γκέρικε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Εμπορίου γιατί πραγματικά θεωρώ ότι και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι εμπορικές συναλλαγές και εγώ είμαι εισηγητής, συντονιστής συγγνώμη, για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και η οικονομία και το εμπόριο χρειάζονται fair play, χρειάζονται ίσους όρους και είναι πάρα πολύ σημαντικό, άκουσα την Επιτροπό που ανέφερε όλους αυτούς τους τομείς. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η συμφωνία αυτή να βασίζεται σε ίσους όρους, σε fair play, στην τήρηση κοινών κανόνων. Μιλάμε λοιπόν για αυτό το fair play και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ισχύσει σε αυτή την εμπορική συμφωνία. Αν θέλετε να κάνουμε κάτι από κοινού, θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Ευχαριστούμε ο κύριος Φερέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Οι διαπραγματεύσεις για αυτές τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου κράτησαν δέκα χρόνια γιατί οι αφρικανικές χώρες αντιστάθηκαν να τις ε, υπογράψουν γιατί δεν προωθείται το εμπόριο διότι οι αφρικανικές χώρες δεν θα έχουν τους πόρους που χρειάζονται και θα αποδιαρθρώσουμε τις αγορές τους. Μιλάμε για μία νέα τάση απεικιοκρατίας αυτό που ε, μας ενδιαφέρει είναι να μην δεχτούν αυτές τις συμφωνίες οι Αφρικανοί ε, με ανοιχτές αγκάλες. Για πολλά χρόνια αυτές οι χώρες έπρεπε να υποστούν τις δικές μας προδιαγραφές και προστάγματα. Όπως φαίνεται από αυτή τη συζήτηση, έμπρακτα δεν σημαίνουν τίποτα αυτές οι συμφωνίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ για ένα λεπτό από την ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που μα εξηγήσατε και πάλι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι στην καρδιά τη στρατηγική εμπορίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ απολύτω. Πώ θα το κάνουμε όμω, ειδού το ερώτημα. Και σε αυτέ τι συμφωνίε θα πρέπει να καταφέρουμε να συμπεριληφθούν με τρόπο αποτελεσματικό ανθρώπινα δικαιώματα που να δείχνουν τα δόντια τους. Ε, η ρήτρα αυτή που αναφέρεται έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να τους τρίζουμε και τα δόντια καμιά φορά. Η παρακολούθηση συχνά δεν απέδωσε, δεν λειτουργήσε ε, προς την κατεύθυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς θα τα εξασφαλίσουμε αυτά, ότι στην Ευρώπη πραγματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα τα βάζουμε στις συμφωνίες που να μην είναι ξεδοντιασμένες και να πίπτει και ράβδος όταν πρόκειται για κυρώσεις. Υπάρχουν προβλήματα εκεί στις συμφωνίες, δεν τα έχουμε καταφέρει, δεν έχουμε κεφάλαιο για την αηφοροανάπτυξη και πιστεύω ότι είναι πρόβλημα αυτό. Πάντως με χαρά θα ακούσω τις προτάσεις σας για το πώς ε, θα ε, έχει κάποια πυγμή αυτή η συμφωνία και θα από ποινές και Ευχαριστώ κύριος Φιέλνε για ένα λεπτό και μισό. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Πρόεδρε. Τώρα λοιπόν οι αριστεροί ε, συχνά ε, συζητούν για αυτές τις συμφωνίες λες και η Ευρώπη προσπαθεί να επιβάλλει και να αναγκάσει τις φτωχές χώρες να δεχτούν τους δικούς μας όρους. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Εμείς διαπραγματευόμαστε και στη συνέχεια υπογράφουμε. Τι είναι αυτά που ακούμε εδώ απόψε. Τους ίδιους αριστερούς που ε, δυσανασχετούν γιατί οι φτωχές χώρες της Αφρικής δεν συμφωνούν μαζί τους. Μα το εμπόριο είναι τρόπος να ε, κρυζωθεί η φτώχεια και να αναπτύσσονται τα κράτη και οι λαοί. Έχω μια ερώτηση Η Αφρική είναι καταδικασμένη να μείνει φτωχή για πάντα. Δεν θέλετε να πλουτίσει. Δεν θέλετε να υπάρχει μεγαλύτερη ευημερία. Τι συμφωνία θέλετε να επιβάλλουμε εμεί του όρου μα ή να ακούμε και του εταίρου μα όταν υπογράφουμε συμφωνίε. Ευχαριστώ. Κύριε Φεραίρα, πήρατε το λόγο προηγουμένω. Δεν μπορώ να σα δώσω τώρα μπλε κάρτα. Για ένα λεπτό, κύριο Μάρτιν. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως προαναφέρθηκε, εγώ ήμουν εισηγητής για ένα συναφές θέμα, το οποίο αποτέλεσε ορόσημο για τη μελλοντική μας ε, πορεία και γι' αυτό εκτός, ε, να, εκτός από το γεγονός ότι μιλάμε για τα περιβαλλοντικά αναφερόμαστε και στο κοτονού. Και όπως ξέρετε, επειδή λίγη η συμφωνία του Κοτονού, δεν ξέρουμε πώς αυτή η ΣΟΕΣ θα ισχύσει στο μέλλον. Θα ήθελα να μας πει η Επιτροπή τι σκέφτεται σε σχέση με τη λήξη του Κοτονού και τις ε, επιπτώσεις της ΣΟΕΣ. Δέχομαι αυτά που είπε η κυρία Σκακέλνερ σε σχέση με την χρηματοδότηση αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ενισχύσουμε τις θέσεις μας και κατά πόσο πραγματικά επιτελείται ε, πρόοδος. Η κυρία Ρένα, στα πλαίσια του Catch the Eye, η πρώτη από τις δύο, από Ευχαριστώ. Δύο, τρεις ερωτήσεις. Ο David Μάρτιν ε, υπέβαλε την πρώτη αναφέρεται στη Συμφωνία του Κοτονού και πώς συμβαδίζει με τη Συμφωνία μας στη Δυτική Αφρική. Ε, μιλάμε για μία νομική υφής ερμηνεία και αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε ποια θα είναι η νομική βάση για, για το διάλογο και τις κυρώσεις. Επίσης, ποιο θα είναι το ευεργέτημα για τις αφρικανικές χώρες, γιατί 12 από τα 16 κράτη ε, εντάσσονται στους στόχους ε, της χιλιετίας. Το South Center ε, έφτασε σε συγκεκριμένα, συγκεκριμένα συμπεράσματα και βλέπουμε ότι ότι οι ζημίες είναι πολύ ψηλότερες από τα κέρδη. Σε σχέση με την Ιγυρία που αντιτάσσεται στεναρά, το καταλαβαίνουμε, γιατί υπάρχει μείωση κατά 7 δις του ΟΕΠ πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε και να απαντήσετε στην Ιγυρία. Ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε σημαντική την ε, διαπραγμάτευση της εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Αλλά βεβαίως πρέπει να υπάρξουν ε, ορισμένες προϋποθέσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχυθεί η συνεργασία των χωρών της περιοχής, διότι μόνο έτσι θα υπάρξει ανάπτυξη. Και υπάρχοντας ανάπτυξη δεν θα έχουμε μεγάλα κύματα οικονομικών μεταναστών οι οποίοι πλέον έρχονται στην ευρώπη. ταυτόχρονα με την περιφερειακή συνεργασία θα έχουμε και εμπέδωση της ειρήνης και έτσι θα μειωθούν οι συγκρούσεις για να έχουμε ένα δεύτερο θετικό αποτέλεσμα να περιοριστούν οι προσφυγικές ροές οι οποίες ξεκινούν και από αυτή την περιοχή και έρχονται στην ευρώπη. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι η παιδική εργασία όπως αναπτύχθηκε είναι πλέον κάτι το οποίο συμβαίνει συνεχώς και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να είμαστε κάθετοι αντίθετα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Κατσιάη. Θα δώσουμε το λόγο και πάλι στην Επίτροπο. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Το εμπόριο είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης και, τη, ε, την διαβίωση γενικότερα. Όπως ξέρετε, οι ΣΟΕΣ δεν είναι συμμετρικές οι συμφωνίες οικονομικής οικονομικής-ετερικής σχέσης και δεν ζητάμε από τις χώρες αυτές να ανοίξουν τις αγορές τους κατά τον ίδιο τρόπο. Ξέρουμε ότι πολλές ε, αγορές είναι πολύ ευάλωτες και θα πρέπει να τις βοηθήσουμε στη διαφοροποίηση. Κυρία Αρένα, συζήτησα με πολλούς φορείς στην Ιγυρία, όπου βρέθηκα πριν από τα Χριστούγεννα και νομίζω ότι θα ευεργετηθούν πάρα πολύ θα υπάρξει διαφοροποίηση της αγοράς τους και θα τους ε, βοηθήσουμε έτσι ώστε να, έχουν, να πληρούν τις προδιαγραφές στο γεωργικό τομέα και θα βοηθήσουμε και στην περιφερειακή τους ολοκλήρωση. Αυτό το νόημα έχουν και οι συμφωνίες ε, οικονομικών εταιρικών σχέσεων. Μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Μίμητσα ασχολούμαστε με την ολοκλήρωση των ΣΟΕΣ. Βεβαίως η βιωσιμότητα είναι ε, θέμα κλειδί και συμφωνώ με την κυρία Κέλλερ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα αλλά προσπαθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουμε με το διάλογο, όχι με τις κυρώσεις. Γιατί αν αρχίσουμε με τις κυρώσεις, τότε δεν θα πληγούν οι αρχές, αλλά ο μέσος πολίτης. Γι' αυτό αρχίζουμε με το διάλογο στα διάφορα φόρα και υπάρχει και η δυνατότητα των κυρώσεων στο τέλος. Αλλά στο μεταξύ έχουμε κάνει πολλά βήματα ως προς τη Συμφωνία Δυτικής Αφρικής. Δεν προωθήσαμε το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης όσο θέλαμε. Γι' αυτό υπάρχει μία ρήτρα για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε περαιτέρω. Αλλά όπως είπα στην εισήγησή μου θα υπάρξει εποπτεία ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντικά, ενέργεια και ούτω καθεξής. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Κύριε Μάρτιν, λίγη συμφωνία του Κοτονού. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Όμως ε, οι διατάξεις ε, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Δεν θα αλλάξουν ε, οι αρχές μας υπάρχει η διαδικασία, και, η διαδικασία εποπτείας και μέσω του κοτόνου ως προς την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό θεωρώ ότι με τις χώρες ΑΚΕ, σήμερα μιλάμε για τη Δυτική Αφρική, αλλά είχαμε διαπραγματεύσεις και με τις χώρες ΑΚΕ. Υπάρχει εταιρική σχέση που θα είναι ευεργετική σε αυτή την περίπτωση για τη Δυτική Αφρική, αλλά και τις χώρες ΑΚΕ, έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη θέσης εργασίας και υποστήριξη της οικογένειας στη χώρα που ζουν μέσα στα πλαίσια της περιφερειακής ολοκλήρωσης που είναι πραγματικά ελληματική. Ευχαριστώ και Επίτροπε,